σε μια ανακοίνωση βάσει του άρθρου 137.2 του κανονισμού έλαβα έτοιμα από την Επιτροπή ΦΑΜ για τη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την κατάσταση των γυναικών Ρωμά. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από πολιτική ομάδα ή το ελάχιστο όριο βουλευτών μέσα σε 24 ώρες, το αίτημα για διαβούλευση θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται